Ξεκινάμε το ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην, στην Κρυμαία και ιδιαίτερα την κατάσταση των Τατάρων. Παράγραφοι προφορική τροπολογία του κυρίου Πλένκοβιτς. Κύριε Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την προφορική τροπολογία για την παράγραφο 7, είναι τεχνικό ζήτημα. Κάτι το οποίο συμφωνήσαμε στις